Θα ήθελα να σας πληροφορήσω επίσης ότι αύριο στις 12 το μεσημέρι στο, στην Ολομέλεια αυτή θα τιμήσουμε τη Σιμών Βέιλ. Άρα μετά από την τιμητική αυτή συνεδρίαση θα γίνει η ψηφοφορία όσοι συμμετάσχουν στην κηδεία που θα λάβει χώρα στο Παρίσι την Τετάρτη στις 10.30 θα μπορέσουν να έχουν δικαιολογημένη αποσία από τις εργασίες του Κοινοβουλίου και της Ολομέλειας. Dichiaro formalmente Άρχεται η συνεδρίαση, επαναλαμβάνεται η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιθυμήσω σε όλους τους συναδέλφους ότι την Παρασκευή λάβαμε μια ιστορική απόφαση. Τελικά η Γερμανία όπως και άλλες χώρες μέλη ενέκρινε, εψήφισε του γάμου μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου. Και αυτό το το Ευρωκοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια έχει δώσει μάχη προ αυτό τον στόχο. Χωρί να έχει βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα το είχε κάνει αυτό η Γερμανία. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προυστ ε, παρόλα. Προυστ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ εντάχει κατά τη σύνοδο αυτή στο Στρασβούργο όπου χτυπάει καρδιά της δημοκρατίας να τιμήσω εξ του ΕΛΚ και της γαλλικής αντιπροσωπείας τη Σιμών Βέιλ η οποία μας εγκατέλειψε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα παραμείνει στη μνήμη μας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν ήταν 16 χρονών πέρασε από το ε, Auschwitz και κατάφερε να επιβιώσει. Συμβάλλει σε μία μεγάλη ελπίδα για όλο τον κόσμο γιατί στάθηκε για τα δικαιώματα των γυναικών και υπέρ της δημοκρατίας. Η Σιμών Βέιλ είχε να αντιμετωπίσει μεγάλα εμπόδια ήταν άνθρωπος της ειρήνης και εργάστηκε σθέναρα για να μπορέσει να συμβάλλει ώστε να μπορέσουν οι πολίτες και οι άνθρωποι να συμβάλλουν στη δημοκρατική διαδικασία. Είχε αναλάβει μεγάλο έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της και οι μεγάλες σειράξεις που επικρατούν στον κόσμο μας δείχνουν τη σημασία της ειρήνης την οποία οφείλουμε στους μεγάλους άνδρες και τις μεγάλες γυναίκες. Η Σιμών Βέιλ ανήκει σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Δυστυχώς χάνουμε αυτά τα σημεία αναφοράς. Αλλά εάν επικρατήσουν τα λόγια, τότε επικρατούν και οι πράξεις η Σιμών Βέιλ μπόρεσε να συνδέσει το λόγο με την αλλαγή. Αύριο θα γίνει μια τιμητική συνεδρίαση για την Σιμών Βέιλ. Θα ήθελα όμως να τονίσω την ε, μεγάλη πορεία αυτής της ε, μεγάλης γυναίκας που μπόρεσε να προωθήσει τη δημοκρατία στο, στην Ολομέλεια και στο Κοινοβούλιο αυτό. Γκίσμπεκ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της ομάδας ε, της Άλντε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συμφωνήσω με τα λόγια σας ε, και να πω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να γίνει αύριο αυτή η τελετή στη μνήμη μιας ε, πάρα πολύ μεγάλης γυναίκας ε, της Σιμον Βέη και ε, επίσης συμμερίζομαι όλους τους Γάλλους αλλά και όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που χαιρετίζουν την γυναίκα αυτή που συμβολίζει τον 20ο αιώνα ένα πολύ σημαντικό μετέχμιο που κλείνει βέβαια με τη ΣΟΑ και βέβαια η φωτεινή προσωπικότητα της Σιμών Βέιλ ε, εκπροσωπεί κάτι σημαντικό και για τον 21ο αιώνα. Ε, μία πολιτικός αλλά μία γυναίκα πάνω απ' όλα η οποία συμφιλίωσε αξίες, απαιτήσεις, ε, διεκδικήσεις με έναν πάρα πολύ έντονο ισχυρό χαρακτήρα που διατέλεσε και πρώτη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη δε χώρα μου έχει εμπνεύσει αξίες οι οποίες ε, βρήκαν μιμητές φυσικά πέραν των εθνικών συνόρων, ε, δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των γυναικών, καθότι ξέρουμε ότι έγραψε πολλά κείμενα σε σχέση με αυτά τα θέματα και ε, χαίρομαι που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα οργανωθεί τελετή στη μνήμη της μεγάλης αυτής γυναικείας προσωπικότητας. και σας ευχαριστούμε εξ ονόματος και της δικής μου πολιτικής ομάδας, στην οποία ανήκει η αλλά και όλων των Γάλλων. Ευχαριστώ. Κυρία Νταλόν Μπονφουά. Euh, Ευχαριστώ πολύ για την απόδοση τιμής ε, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με τους προλαλήσατε συναδέλφους ε, Γκρισμπέκ και Προύστα. Ε, Σιμών Βέιγε με όλη της την πολιτική σταδιοδρομία κατάφερε να συσπυρώσει και έκανε τα μάλα για την Ευρώπη και για την αναγνώριση της Ευρώπης. Στη Γαλλία έκανε όμως ε, τα μάλα και για τα δικαιώματα των γυναικών. Ιδίω δε σε θέματα άμβλωσης ε, που πλέον είναι νόμιμη ε, και αυτό ήταν μια μάχη πάρα πολύ σκληρή που έδωσε η Σιμουν Βέλ, και που δώσαμε όλοι μας και συνεχίζουμε να δίνουμε οι σοσιαλιστές ε, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε τιμώντα τη μνήμη της ε, ώστε να μην είναι επιματέο αγώνα, να μην ε, λήξει και να μπορούν να ωφεληθούν όλοι οι Ευρωπαίοι από το έργο της μεγάλης αυτής γυναίκας της οποίας θα τιμήσουμε τη μνήμη. Ευχαριστώ. Πράγματι, η Σιμών Βέιλ άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό τιμούμε τη μνήμη της. Λούνατσεκ. Και εγώ θα ήθελα εξ ονόματος των Πρασίνων να σας ευχαριστήσω γιατί τιμάτε τη μνήμη της Σιμών Βέιλ ήταν μια πολύ σημαντική μορφή για τα δικαιώματα των γυναικών στη Γαλλία αλλά και σύμβολο για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και θα ήθελα να την τιμήσουμε για το έργο της υπέρ της Ευρώπης. Η κυρία Τόγια ζήτησε το λόγο, αλλά σας υπενθυμίζω ότι αύριο θα αποδοθούν τιμές στην ε, κυρία Βέιλ, στην Σιμών Βέιλ και γι' αυτό δεν πρέπει να επεκταθούμε εδώ. Θα ήθελα να πω ότι πολλές φορές πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη σημασία σε χώρες που αντιμετωπίζουν ε, μεγάλα θέματα στον τομέα της μετανάστευσης. Ε, δυστυχώς το τελευταίο διήμερο έφτασαν 12.000 στις ακτές μας και την επομένη 5.000. Και λέω δυστυχώς γιατί φυσικά θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, αλλά θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη και ενωτικό πνεύμα. Γιατί εμείς καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες. Η Ιταλία και η Ελλάδα πρέπει να ε, τύχουν της βοηθείας των υπολείπων μέσα στα πλαίσια της αλληλεγγύης. Μιλήσαμε για τη Σιμών Βέιλ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επιδείξουμε ενωτικό πνεύμα όπως επιδείκνει και η Σιμών Βέιλ σε πλήστες όσες περιστάσεις. Κυρία Τόγια, θα συζητηθεί και το ζήτημα αυτό μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της Εσθονικής Προεδρίας. Μίλησα με τον Πρωθυπουργό Ράτας, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι το μεταναστευτικό είναι ύψης της σημασίας. Τα πρακτικά έχουν διανεμηθεί, τα πρακτικά του Ινίου υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι, άρα εγκρίνονται τα πρακτικά. Μετά τον διορισμό του κυρίου Ιαν Ντάνκα